Κύριοι, ε, αύριο θα συνεδριάσουμε Τετάρτη ε, στις 9 Οκτωβρίου από τις 9 ε, μέχρι τις 2 και από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ. Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε και είναι στην διάθεσή σας.